Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μου με ενημέρωσαν ότι έχει αρθεί η ασυλία του κυρίου Πόλσακ και έτσι λύγει και η διαδικασία άρσης